Mes chers collègues, bonjour. καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Monsieur Robert Zille, prenez votre temps. Hein. Ναι, ναι, όχι, μην βιάζεστε. Σιγά σιγά, καθίστε. Très bien. Πολύ ωραία. Καλημέρα σα. Είναι Πέμπτη, είναι η τελευταία μέρα του Στρασβούργου, αλλά θα τα πάμε όλα καλά. Λοιπόν, σχέδιο τη διάταξη εγκρίνεται αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Υπάρχουν αντιρρήσει, Όχι. Ε, Ανακοινώσει τη Προέδρου. Θα ήθελα να σα ε, ενημερώσω ότι ο κύριος Έρτογκ που είναι μέλος των σοσιαλιστών που μόλις ορίστηκε αντιπρόεδρος της ομάδας του συγχαρητήρια κύριε Ερτούγκ και ο συντονιστής Άρα δυστυχώς δεν μπορείτε να είστε πια και συντονιστής. Και έχω την τύχη ο κύριος Διέρεσον να γίνει συντονιστής του σοσιαλιστικής ομάδας. Συγχαρητήρια και σε εσά. Και τώρα που τα γνωρίζετε όλα αυτά, θα ξεκινήσουμε αυτό που όλοι περιμένετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως το γνωρίζετε, οι συντονιστές της Επιτροπής μας δεν θέλησαν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει στο Κοινοβούλιο με τις τρεις προτάσεις της δέσμης ε, κινητικότητα, αλλά η ομάδα ECR ε αμφισβήτησε την απόφαση αυτή των συντονιστών, οπότε σήμερα πρέπει να ε, λάβουμε μία απόφαση με ψηφοφορία. Γι' αυτό αμέσως θα ψηφίσουμε για αυτό το ζήτημα. Κύριε Ζηλέ, θέλετε να πάρετε το λόγο πριν να εξηγήσω πώς θα γίνει. Επειδή είστε εσείς, σας δίνω το λόγο. Εξ ονόματος του ECR, θα ήθελα να ζητήσω να έχω γίνει ονομαστική ψηφοφορία γιατί χρειάζεται συγκεκριμένος αριθμός μελών. Μάλιστα. Ο κύριος Ζήλε θέλει λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία να γίνει. Μάλιστα. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της πρότασης. Πρέπει να σηκωθείτε. Εντάξει, μπορείτε να ξανακαθίσετε. Για τους νεοφυχθέντες, ο κανόνας είναι απλός. Έχει κάνει το δικαίωμα να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία εφόσον πάνω από 10 βουλευτές το ζητήσουν. Κάποιος μου έσβησε το μικρόφωνο μου. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάνω από 10. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Προσέξτε. Η ερώτηση για την οποία ψηφίζουμε είναι η εξής. Θα τη βρείτε και στον κατάλογο ψηφοφορία σας, αλλά σας το θυμίζω. Επιθυμείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει στο Κοινοβούλιο και να επανεπιβάλλει στις τρεις προτάσεις της δέσμης ε, κινητικότητας. Θα ήθελα να είμαι σαφής για αυτό το θέμα. Δεν θα αρχίσουμε συζήτηση, γιατί Κύριε Ντελή, ναι, κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, δεν υπάρχουν ενδείξεις στα κουμπιά και πολλοί συνάδελφοι δεν ξέρουν ποιο κουμπί είναι υπέρ, ποιο είναι κατά και ποιο είναι αποχή. Μήπως μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμή. Κύριε Ντελή, Monsieur je réponds directement à votre question. Κύριε Ντέλη, θα απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σας. Κύριε Ρόμπερτ Ζήλε, ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, ούτως ή άλλως γίνεται μια δοκιμή, για, θα σας εξηγήσω στους καινούριου πώς λειτουργεί Να σας εξηγήσω λοιπόν πώς λειτουργούν όλα αυτά. Η κυρία Γραπίνη. Ναι, ναι, θα είμαι πολύ σύντομη. Κυρία Πρόεδρε, Έχουμε αρκετού νέου συναδέλφου. σω πριν από την ψηφοφορία θα έπρεπε να του προσφέρουμε μια εξήγηση όσοι επιθυμούν να λάβουν το λόγο για αυτή την υπόθεση, να του εξηγήσουμε περί τίνο πρόκειται. Κυρία Γκραπίνη, η απάντησή μου είναι καθαρή όχι. Δεν θα αρχίσουμε συζήτηση για τη δέσμη, για την κινητικότητα. Εδώ σήμερα το πρωί είστε υπεύθυνοι. Η ερώτηση είναι μία. Θέλετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει και να επαναποβάλει στο Κοινοβούλιο τις τρεις προτάσεις της δέσμης κινητικότητα. Εάν επιθυμείτε η Κομισιόν να κληθεί σε διαβούλευση εκ νέου λοιπόν, θα απαντήσετε ναι και ο η νομοθετική διαδικασία για αυτή τη δέσμη ε, μηδενίζεται και ξαναρχίζουμε αυτού και από την αρχή. Περί αυτού πρόκειται. Η δεύτερη πιθανή απάντηση, εάν επιθυμείτε να ακολουθήσετε την απόφαση των συντονιστών της Επιτροπής Τραν, θα απαντήσετε όχι στην ερώτηση και άρα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα δέσμη κινητικότητας και οι εργασίες θα συνεχιστούν από εκεί που βρίσκονταν το τέλος της περασμένης θητείας. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Καταλάβατε όλοι. Ναι, ο κύριος Μαρινέσκου. Ναι, η ερώτηση είναι πολύ σαφής, αλλά... Δεν πρέπει να πείτε ότι ξαναρχίζουμε από το μηδέν, γιατί η Κομισιόν μπορεί να αρνηθεί, μπορεί να φέρει νέο κείμενο ή να στείλει συμβιβαστικό. Ναι, ωραία. Θα το διορθώσω. Μάλιστα. Θα το, Όχι. Οι βουλευτές εδώ δεν είναι ανόητοι. Αντίθετα. Ναι, όταν λέω θα ξεκινήσουμε από το 0, εννοώ από το 0 του κειμένου. Και, και όχι... Λοιπόν, αρχίζουμε την ψηφοφορία για να δούμε αν έχουμε απαρτία. Ε, άρχεται η ψηφοφορία δοκιμή για να δούμε αν έχουμε απαρτία πρώτα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ε, στο ΕΛΚ ψηφίζουν τέσσερις παραπάνω. Πέντε τώρα παραπάνω. Υπάρχουν υπερβολικά πολλοί από το ΕΛΚ. Ένας τώρα παραπάνω από τον αριθμό που πρέπει. Αποφασίστε ποιος δεν θα ψηφίσει. άντε. Ακόμα υπάρχει ένας Συμφωνήστε μεταξύ σας. Bon, allez. Bon, et le PP. Il y en a un. Ακόμα έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ. Το λέει το μηχάνημα. Εμπιστευτείτε το μηχάνημα. Κύριε Μαρινέσκου, μην κοιτάτε τον κύριο Ρικέ, γιατί δεν είναι στην ίδια πολιτική ομάδα με εσάς. now it's Allez. Et désormais... Ωραία. Οπότε, κηρύσω την έναρξη της ψηφοφορίας για το ζήτημα αυτό επίσημα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε παρακαλώ. Le vote Πέρα τη ψηφοφορία. Η πρόταση απορρίπτεται. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας λοιπόν. Τελειώσαμε. Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα. Την τρίτη δηλαδή που μας έρχεται από τις 9 το πρωί. Κυρίσω τη λήξη της συνεδρίασης.